Λοιπόν, αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Ντόλτεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Λόρδος Έμραϊ βοήθησε έτσι ώστε η Europol να γίνει ένα σημείο ανταλλαγής πληροφοριών πολύ πολύτιμο ανάμεσα στις νομικές αρχές. Σήμερα κάναμε ένα βήμα ακόμα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος με την ε, βοήθεια εμπειρογνωμόνων και των ευρωβουλευτών. Η Europol, ε, η, αυτή, αυτή η ενότητα της, ε, αυτή η μονάδα της Europol άρχισε να λειτουργεί πριν από ένα χρόνο και έχει βοηθήσει πάρα πολύ ήδη πάνω από 700 ε, 700 συστήματα ε, διαγραφής πληροφοριών έγραφε το πρώτο, έλαβε το πρώτο εξάμεινο. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση θα βοηθήσει τη Europol να προχωρήσει και να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και στο μέλλον. Γι' αυτό την υποστήριξα. Παρακαλώ συνάδελφοι, λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η κυρία Μορβάη. Mrs. Morvai. europol Η Europol είναι μια ε, υπηρεσία υπεύθυνη και αρμόδια για την αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη. Ε, έχει ως αποστολή να καταπολεμάει το έγκλημα και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από τους πολίτες. Ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας, ε, λαθρεμπόριο ανθρώπων κλπ. είναι μέσα στην αποστολή της. Δεν θα ήταν λοιπόν ώρα, δεν έχει έρθει ο χρόνος να έρχονται εδώ οι υπεύθυνοι της Europol και να μας εξηγούν και να μας εξηγήσουν τι έχουν κάνει με τα χρήματα που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Πολλοί πολίτες μου στέλνουν επιστολές που με ρωτάνε γιατί σε τι χρησιμεύει η Europol, γιατί δεν κατάφερε να αποφύγουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τους λαθρεμ, το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Τι μπορούν να μας πούν ότι έκαναν για να καταπολεμήσουν τα διεθνή δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Σε τι χρησιμεύουν τα λεφτά που τους δίνουμε. době má smysl posílit pravomoce europolu nejsem příznivcem zřizování nových úřadů osobně nepodporuji zřízení například nového. Δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων ε, οργάνων, ε, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπόλ στο μέλλον θα πρέπει να δίνει στις διάφορες, στα διάφορα, στις διάφορες ε, αστυνομικές δυνάμεις πληροφορίες για τις τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να έχει πληροφορίες ε, από τα διάφορα κράτη-μέλη. Οπότε συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Γιατί ενισχύει την ειδική μονάδα της Europol για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Mulțumesc. Un mandat mai puternic al Europol este πιο ισχυρή εντολή προς την Europol αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών μας και είναι υποχρεωτικό η Europol να έχει μια σύγχρονη βάση δεδομένων και να προβαίνει σε σύγχρονη διαχείριση των δεδομένων. Αυτό είναι νομικό προαπαιτούμενο, αφορά και ιδιωτικού φορεί και διεθνεί οργανισμού. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο παντού. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα αν δεν υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στου εποπτικού φορεί ε, και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω ε, διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί ε, και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στέλνουν τι απαραίτητε πληροφορίες ε, ας πούμε στην Τράπεζα Δεδομένων του Σέγκεν που σημαίνει ότι η Τράπεζα Δεδομένων του Σέγγεν δεν περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν ανθρώπους που θα μπορούσαν να επιτεθούν στην Ευρώπη ή <clears throat> να έχουν ενταχθεί σε τζιχαντιστικές ομάδες. Καλό λοιπόν τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες να στέλνουν τα δεδομένα τους στην Τράπεζα Δεδομένων του Σέγγεν. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπαν, λέει ο ότι το κρίμα δεν αφορά τα διεθνή σύνορα και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κράτη-μέλη έχουν συνεργαστεί. Έχουμε την Ίντερπολ, έχουμε συμφωνίες απέλασης. Ε, όλα αυτά είναι εργαλεία ε, τα οποία ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτή η Europol. Όπως υπόθηκε πολύ σωστά, όταν η Europol πρώτο συστήθηκε ήταν για να υπάρχει μια ομοσπονδιακή αστυνομία. Ένα είδος ευρωπαϊκού FBI. Και για μας αυτή ήταν η επιλογή ανάμεσα στην ε, σύνδεση και την απορρόφηση, ε, συμμαχία και ταύτιση, συνεργασία και εξαναγκασμός. Ευχαριστούμε. Τώρα κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, η ρύθμιση που προτείνει το Συμβούλιο θα βελτιώσει το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί καθημερινά η Europol. Το έγγραφο αυτό λοιπόν θα αρχίσει να ισχύει από τον Μάιο του 2017. Τότε θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η υπηρεσία της Europol. Υπάρχουν πολλοί, πολλές δυνατότητες για βελτίωση της απαταλισματικότητας της Europol και επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούν να αξιολογήσουν το έργο της Europol εφ' μέσω μιας ειδικής ομάδας εργασίας. Ο προπολογισμό θα αυξηθεί επίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άρνοτ, λέει Ευχαριστώ. Όλοι θέλουμε συνεργασία, όλοι θέλουμε αποτελεσματικότητα, όλοι θέλουμε να δουλεύουμε μαζί με την Europol και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να δουλεύει και με το 5i και με τα δίκτυα τα σχετικά. Και περισσότερη διαφάνεια από την Europol. Η εκστρατεία στον Ηνωμένο Βασίλειο λέει μεταξύ άλλων ότι άμα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται η ασφάλειά μας. Σκότ Γιάρτ είπε ότι το ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθάει να αντιμετωπίσουμε απειλές από το εξωτερικό. Και ο Μάκρετ είπε ότι οι σχέσεις ανταλλαγής πληροφοριών είναι με ατομικά κράτη-μέλη και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Άρα λοιπόν, άμα θέλουμε να είμαστε παρόντα στο διεθνές επίπεδο, φυσικά και πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλες χώρες μέλη. Αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε τέλεια να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να διασφαλίζουμε την εθνική μας προστασία χωρίς να πρέπει να είμαστε ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταψήφισα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μαουλού. Ε, σωστή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε. Το να ενισχυθεί η Europol σημαίνει ότι ενισχύουμε την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να ακολουθεί ένα κριτήριο το οποίο θα είναι άκαμπτο και αυτό για να μπορούμε να αγγιόμεθα την ε, νέα μορφή ομοιομορφία, την συλλογή πληροφοριών ε, και το θέμα τη πρόσδευαση στο ε, διαδίκτυο. Γιατί από εκεί προσελητίζουν νέου μετά του εντάσσουν σε τρομοκρατία είναι λοιπόν ε, μια πολύ θετική προσέγγιση. Εγώ υπερψήφισα και είμαι υπερήφανο που το Κοινοβούλιο ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Πολτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δεν έχουν σύνορα. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεργαζόμαστε επιτυχημένα. Η Europol, ε, παρόλες τις κάποιες αδυναμίες της, ε, έχει κερδίσει το σεβασμό των πολιτών μας. Είναι ένας οργανισμός που θα πρέπει να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο την ε, αστυνομική συνεργασία. Στήριξα λοιπόν αυτή την έκθεση. Ε, δεν, ο στόχος δεν είναι η δημιουργία μιας ομοσπονδιακής αστυνομίας, αλλά χρειάζεται να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας. Και η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένου κανόνες. Ε, η έκθεση αυτή δεν αποφεύγει να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ. Κέλλη. Ε, Όπως και η περισσότεροι ευρωβουλευτές και εγώ υπερψήφισα την σύσταση αυτή. Δίνουμε τώρα με αυτόν τον τρόπο στην Europol τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αυτό το κείμενο θα πρέπει να το δούμε με, παράλληλα με την ψηφοφορία που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες για τα μητρώα επιβατών. Ε, κάνουμε λοιπόν πρόοδο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αυτό είναι πράγματι πολύ καλό. Οι πολίτες μας, οι άνθρωποι μας ε, γνωρίζουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο ασφαλής στο μέλλον. Προσθέτουμε 2,1 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό της ε, Europol και είναι ένα ποσό που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στην δεύτερη ανάγνωση, σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης Σεσίλια Βίλκστρομ. Η κυρία Μορβάη έχει το λόγο πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Βίλκστρομ απέρριψε χωρίς να δικαιολογήσει το αίτημα που είχε να κάνει με τα δάνεια σε ξένο νόμισμα. Κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τους Ούγκρους ερευνητές και φοιτητές. Η μετανάστευση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το... η ζήτηση ανθρωπίνου δυναμικού πρέπει να είμαστε σε θέση να υποδεχόμαστε καλύτερα τους φοιτητές και ερευνητές που μας έρχονται από τρίτες χώρες. Γιατί για μας είναι κάτι που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρειάζεται αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις. Κυρία Βίλστρομ, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τους πανεπιστημιακούς ερευνητές Ούγγρους πριν να γράφετε πράγματα όπως έχετε γράψει εδώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Η ανταλλαγή φοιτητών, οι ερευνητές, η απασχόληση εσωτερικών άμυστων βοηθών, η επιπληρωμή. Είναι πράγματα που όντως πρέπει να προσέξουμε και αυτό ακριβώς έχουμε κάνει τώρα. Η κινητικότητα μεταξύ των νέων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και για να ενισχύσουμε τα προσόντα του εργατικού μας δυναμικού. Αν έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, τότε το ανθρώπινο δυναμικό θα έχει ψηλότερα προσόντα. Άρα η δουλειά που θα κάνει θα είναι καλύτερη και θα εξελιχθεί και καλύτερα η κοινωνία έτσι. Ανοίγοντας λοιπόν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικόους τρίτων χωρών, εξακολουθούμε να πρέπει να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφύγουμε εκείνους οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη τάχα μου για να σπουδάσουν ή για να δουλέψουν, αλλά φέρουν και τον εξτρεμισμό μαζί τους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ποσπίσιλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, στηρίζω το σχέδιο αυτό, το κείμενο για τον ε, εξή λόγο. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να στηρίξουμε την κινητικότητα των νέων, είτε αυτοί είναι φοιτητέ είτε ερευνητέ. Τη στιγμή όμω που προσπαθούμε να βάλουμε κανόνε, ενιαίου κανόνε, ομοιόμορφου, προκειμένου οι φοιτητέ, οι ερευνητέ από τρίτε χώρε να έρχονται και να δουλεύουν ή να σπουδάζουν στι χώρε μα, συγχρόνω, που το βρίσκω θετικό, συγχρόνω Ευρωπαίοι φεύγουν από την ε, Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιώσουμε και την ποιότητα των ε, σπουδών και της έρευνας μέσα στην Ευρώπη για να κρατήσουμε και τους δικούς μας και για να προσελκύσουμε και ακόμα περισσότερους απ' έξω γιατί μόνο τότε μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες μας και έτσι να ενισχυθεί πράγματι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι σε άλλες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία κλπ. Ευχαριστούμε κύριο Χάναν. Ευχαριστώ. Το θέμα της ε, μετανάστευσης έχει οδηγήσει σε τραγωδίες. Έχουν καταργηθεί σύνορα και κρατάμε μόνο τα εξωτερικά. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια νέα χώρα και να έχει μόνο ένα σύνορο και όχι εσωτερικά σύνορα, εντάξει. Αλλά πληρώνουμε με την κρίση μια τέτοια ιδέα, με το δόγμα αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές συνέπειες, όπως και το ευρώ, το οποίο την ε, ολοκλήρωση δεν την πετυχαίνει. Δηλαδή, το δίλημα της 23ης Ιουνίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακριβώ αυτό. Επειδή εμείς έχουμε το δικό μας νόμισμα, επειδή έχουμε τα δικά μας διαβατήρια, μπορούμε να κάνουμε τις δικές μας επιλογές απέναντι σε εμά και απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε, Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε χρόνο εκατομμύρια αλλοδαποί φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σπουδάσουν, ε, να ερευνήσουν για ε, λόγους εθελοντισμού κλπ. Και αυτό είναι πολύ καλό. Η καινούργια οδηγία έχει στόχο την βελτίωση της νομοθεσίας που τους αφορά και τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες για τον έλεγχο της εισόδου αυτών των ατόμων ε, και αυτό είναι επίση καλό. Το Συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση της Κομισιόν βέβαια σε ό,τι αφορά τους φοιτητέ και την εργασία τους και τους επιτρέπει να εργαστούν 15 ώρες ε, για τους ανθρώπους που είναι σε μαθητεία ε, υπάρχει ένα όριο 6, ένα ελάχιστο όριο 6 μηνών ε, με ένα μέγιστο όριο 6 μηνών που μπορεί βέβαια να το παρατείνει το κράτος. Ευχαριστώ pane předsedající samozřejmě posilování mobility. ο eh, Η ενίσχυση της ε, κινητικότητας των νέων, οι ανταλλαγέ, ε, οι νέοι σε μαθητεία, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθούν. Τώρα υπάρχουν θέματα ασφάλειας βέβαια, και τα οποία δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε χρειάζεται να ελέγχονται επαρκώ όσοι φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω τα θέματα ασφάλεια δεν μπορούν να επισκιάσουν όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα. Κίνδυνοι υφίστανται, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε τις επαφές μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων κλπ. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Θα πρέπει να το αποφύγουμε γιατί οι ανταλλαγές βελτιώνουν την ποιότητα της επιστήμης, ε, ε, προωθούν την ε, ευρωπαϊκή επιστήμη κλπ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πάλι λοιπόν πιστεύω ότι είναι θαυμάσιες οι συστάσεις αυτές και το μόνο που μπορούν να επιφέρουν είναι καλό όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βέβαια πάρα πολλά για πολλά χρόνια για τις αναπτυσσόμενες χώρες, του έχει προσφέρει κάθε μορφής βοήθεια, αλλά Πιστεύω ότι τώρα πια πρέπει να εφαρμόσουμε αυτές τις ε, συστάσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι που έχουν δεξιότητες αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα στις χώρες τους να ε, χρησιμοποιήσουν και να αξιολογηθούν αυτές οι δεξιότητές τους αυτοί να μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασχοληθούν με την έρευνα, με τον εθελοντισμό και εάν παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν ένα σημαντικό δυναμικό προς εκμετάλλευση και όταν πια θα επιστρέψουν στις ε, πατρίδες τους ε, θα έχουν ε, εμπειρία που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τότε πια στις επιχειρήσεις της πατρίδας τους. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος που αφορά στην επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής. Η κυρία Μόρβαη. Ευχαριστώ. Τα, τα ταμεία πολιτικής ε, συνοχής έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και η επιτάχυνση υλοποίηση πολιτικής συνοχής είναι αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Προτείνονται λύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω χρήσεως αυτών των ταμείων. Το μόνο που μου άρεσε ήταν η ανάλυση Πολύ συχνά οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν πολύ λίγες πληροφορίες ε, για τις δυνατότητες που έχουν ε, στη διάθεσή τους και αυτό είναι σημαντικό να βελτιωθεί. Το πώς δηλαδή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τα, τις διάφορες αναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν τα χρήματα αυτών των ταμείων είναι γνωστό πως δεν φτάνουν ε, καθ' ολοκληρία στους δικαιούχους τους, πολύ συχνά χάνονται σε ατραπούς διαφθοράς. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται και διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ περιφερειών. Ευχαριστώ κύριο Σόγκορ. Η πολιτική συνοχή έχει ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερων επιτυγμένων περιοχών. οι διάφορες ε, περιφέρειες ε, θα πρέπει να μπορούν να ανταγωνίζονται επίσης όρις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αν θέλουμε να αναζωογονήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαφορά ε, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στις υποδομές μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική συνοχής δεν είναι φιλανθρωπία. Παρά όλα αυτά μερικές φορές επικρατεί σύγχυση για αυτό το θέμα. Χωρίς μια επαρκή πολιτική συνοχή, ε, οι υποδομές ε, και η ευημερία στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές θα βελτιωθούν με πιο αργό ρυθμό από ό,τι στις υπόλοιπες. Και αυτό θα δημιουργήσει, θα αυξήσει την απογοήτευση που υφίσταται. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε την πολιτική συνοχή και να δούμε ποια θα είναι και μετά το 2020, να αξιολογήσουμε ε, ποια, είναι η, ε, ποια είναι τα αποτελέσματά της και στα παλιά κράτη-μέλη. Λόπες Μπερμέχου. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να αποσυνδέουμε τη συζήτηση για την περιφερειακή συνοχή από ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο. Δεν μπορεί να ζητάμε ελαστικότητα από τα δημόσια κονδύλια, να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα που παρέουν από τη λιτότητα και συγχρόνως να επιμένουμε σε νέες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που είναι και η κύρια αιτία των αυξανόμενων ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεγελιόμαστε. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνδέονται όλο και περισσότερο με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες από τις ιδιωτικοποίησεις και το, την ελευθέρωση της αγοράς πάνω στους πολίτες. Δεν πρέπει αυτό να είναι η προτεραιότητά μας, οι ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Όχι. Αντίθετα, πρέπει να αποτελεί η πολιτική μας έναν πόλο για μια διαφορετική παραγωγικότητα οι χώρες μέλη, οι περιφέρειες πρέπει να δούμε πώς έχουν δαπανίσει τα κονδύλια. Το έχουν κάνει συνήθως χωρίς να λάβουν υπόψη τους τον κοινωνικό διάλογο και τους κοινωνικούς εταίρους και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Στην ε, πολιτική συνοχής έχουμε 360 δισεκατομμύρια από το 2014 μέχρι το 2020 που είναι το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Στην προηγούμενη περίοδο υπήρχαν ένα σωρό προβλήματα με τη χρήση των κονδυλίων αυτών από τις χώρες μέλη, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ικανοτήτων από την τοπική αυτοδίκηση και από τους δικαιούχους γενικότερα των κονδυλίων αυτών, συχνά εξαιτία γραφειοκρατικών εμποδίων ή εξαιτία Εξαιτίας ε, διαδικασιών, ε, διαγωνισμών που κράταγαν ε, μεγάλα χρονικά διαστήματα εξαιτίας διαφθοράς ή απλώς ανικανότητας αυτών που διαχειρίζονται αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό και χαιρόμαστε για την διαδικασία στην οποία μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει όλες αυτές τις διαδικασίες για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Απλοποίηση χρειάζεται πρώτα και στη συνέχεια διαφάνεια. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος ζητάει τι, πόσο κοστίζει και πόσο καλά λειτουργεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάμεκίνης. Ευχαριστώ πολύ. Η πολιτική συνοχή, όπως γνωρίζουμε, είναι μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, χώρες, όπως και η δικιά μου η Λετωνία, για παράδειγμα, όπου κάθε χρόνο δεν ζητάει τέτοια κονδύλια και αυτό οφείλεται σε γραφειοκρατικά εμπόδια και στην έλλειψη ενημέρωσης. Έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη πολλών κλάδων στη χώρα μου. Γι' αυτό λοιπόν, με εκείνους οι οποίοι ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες στους δικαιούχους για τις δυνατότητες, για τις ευκαιρίες που έχουν. Πρέπει να κάνουμε πιο λογικό το σύστημα. Να υπάρχει ένας, ένα καλό χρονικό διάστημα σχεδιασμού και η κάθε χώρα να μπορεί να παίρνει τα κονδύλια που της αναλογούν και αν δεν τα καταφέρει την επόμενη περίοδο να πάρει λιγότερα κονδύλια. Αυτό θα ήταν το σωστό. Ευχαριστούμε ο κύριος Πόλσακ. Ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχή η συνοχής υποφέρει από διάφορες ασθένειες, υπερβολική γραφειοκρατία, διοίκηση. Σίγουρα η πολιτική συνοχής δεν επικεντρώνεται επαρκώς στα αποτελέσματα. Δεν αξιολογείται βάσει αποτελεσμάτων. Όλες αυτές οι ασθένειες είναι γνωστές και αντισταθμίζονται από τις ε, παροχές η Ευρώπη θα μπορούσε να ήταν περήφανη αν δεν υπήρχαν διαφορές κατακαιρματισμός ανάμεσα στις περιφέρειες. Άρα λοιπόν είναι μια πολιτική που βοηθάει τις περιφέρειες παρά τις ασθένειες από τις οποίες υποφέρει. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μπορέσει να βρει μια συνταγή για να απλοποιήσουμε την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα παρακολουθήσω από κοντά τα αποτελέσματα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Etheridge. Η στις δημοτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εργατικοί και οι συντηρητικοί λένε δεν έχουμε λεφτά ούτε για θέατρο, ούτε για μουσεία, ούτε για μέτρα οδικής ασφάλειας κλπ. Και παρόλα αυτά αυτοί οι ίδιοι, αυτές οι ίδιες ε, πολιτικές δυνάμεις στηρίζουν τη σπατάληση εκατομμυρίων ε, ευρώ από τα χρήματα των φορολογημένων ε, για τα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ντροπή. Ε, ε, στο σπίτι, ε, στη χώρα μας κλαίνε ότι δεν έχουν λεφτά και από την άλλη μεριά σπαταλούν τα χρήματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι κατά της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης των Ταμείων Συνοχής και είμαι κατά των Ταμείων Συνοχής και θα παραμείνω αν θέλει ο Θεός κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπαταλάμε αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των, των Βρετανών πολιτών. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτή τη σύσταση. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική πολιτική, η πολιτική συνοχή, εξαιρετική ιδέα. 33 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για αυτή την περίοδο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω θα συνεχιστεί και μετά το τέλος αυτής της περίοδου. Γιατί βλέπουμε το δυναμικό που έχει αυτή η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε πως μέσω της πολιτικής συνοχής οι πιο πλούσιες χώρες βοηθούν τις πιο φτωχέ. Όταν ε, εμείς γίναμε μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν πολύ φτωχή χώρα, λάβαμε χρηματοδότηση από την Ένωση και παραδοσιακά ε, και σταδιακά αναπτυχθήκαμε και είμαστε από τι πιο πλούσιες πλέον. Χάρη σε αυτά τα κονδύλια που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ όμως για την ανάγκη να κάνουμε περισσότερο γνωστό το έργο της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. E Thank you very much. Uh, ședința se suspendă până la orele 15. Ε, διακόπτουμε για μέχρι τις 3.